Pan Przewodniczący! Good morning. Witam koleżanki, kolegów. Καλημέρα, καλώ ήρθατε όλοι. Συνεχίζεται η σύνοδός μας. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη ε, η έκθεση του κυρίου Βινταλκάδρας όσον αφορά τον ασφαλή αφοδιασμό με αέριο. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και πολλά χρόνια